Αρχίζει και πάλι η συνεδρίαση, τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης και τα εγκεκριμένα κείμενα έχουν ήδη διανεμηθεί. Θα ήθελα να γνωρίζω εάν υπάρχουν παρατηρήσεις. Δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, συνεπώς θεωρώ ότι έχουν εγκριθεί τα πρακτικά. Περνάμε στην παρουσίαση εκ μέρους του Συμβουλίου της θέσης του σχετικά με το σχέδιο Γενικού Προπολογισμού Οικονομικό έτος 2014. Θα ήθελα να ενημερώσω ότι για την συζήτηση δεν προβλέπεται η διαδικασία Eye, ούτε θα γίνουν δεκτές οι μπλε κάρτες. Θα ήθελα καταρχάς να δώσω το λόγο στον κύριο Αλτζιμάντας Ριμκουνάς, εξ ονόματος του Συμβουλίου. Ε, thank you, Mr. President. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι τιμή μου να σας παρουσιάσω σήμερα τις θέσεις του Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο Γενικού Προπολογισμού για το Οικονομικό Έτος 2014. Ο πρώτος ετήσιος προϋπολογισμός υπό το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο διοθετήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, ευθύ εξ αρχή θα ήθελα να σα διαβεβαιώσω ότι το Συμβούλιο είναι έτοιμο να συνεργαστεί και με το Κοινοβούλιο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι ερχόμενε εβδομάδε και μήνε για να μπορέσει να διασφαλίσει μια συμφωνία για έναν ρεαλιστικό και εξισορροπημένο προϋπολογισμό. Είναι αναγκαία η στενή και αποδοτική συνεργασία. Το Συμβούλιο από μέρου του είναι διατεθειμένο να εργαστεί επικοδομητικά και στα πλαίσια συμβιβασμού και με πνεύμα συμβιβασμού. Ο τρίλογος για τον προπολογισμό που έλαβε χώρα την προηγούμενη εβδομάδα στις 3 Σεπτεμβρίου ήταν θετικός και ιδιαίτερα ενθαρρυντικός. Με χαροποίησε ιδιαίτερα το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησε ως προς την προτεραιότητα που αποδίδουμε σε προγράμματα και δράσεις που υποστηρίζουν την απασχόληση και την ανάπτυξη. Θα ήθελα να τονίσω ως προς αυτό το θέμα ότι το Συμβούλιο σε γενικές γραμμές δέχεται τα ποσά που προτείνονται από την Επιτροπή στο Σχέδιο Προπολισμού 2014 για όλες τις λειτουργικές δαπάνες που έχουν σχέση με προγράμματα υπό το νέο πολιτιές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα επιθυμούσα να αναφέρω ότι όλες ε, οι μειώσεις που προτίθηκαν από το Συμβούλιο βασίζονται σε μια λεπτομερή ανάλυση των, της ενδεκόμενης εφαρμογής μεμονωμένων προγραμμάτων και δράσεων και ότι δεν υπάρχει γενική ε, προσέγγιση ή μη αιτολογημένε περικοπέ. Η μη ειτολογημενε περικοπε η αποψη του Συμβουλίου ω προ το σχέδιο γενικού προπολογισμού υπό το νέο πολιετέ δημοσιονομικό πέσιο προβλέπει 142,2 δισεκατομμύρια σε δεσμεύσει και 135 δισεκατομμύρια ευρώ σε πληρωμέ. Υποστηρίχθηκε από την πλειοψηφία των χωρών μελών. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σα σε τρία σημαντικά στοιχεία που απαρτίζουν τη βάση της άποψης της θέσης του Συμβουλίου. Καταρχάς το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει προτεραιότητα στα προγράμματα και δράσει που είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να ξεκινήσει η Ευρώπη την βιώσιμη ανάπτυξη θέσεων εργασίας αλλά και να ξεκινήσει στον τομέα του εράσμου, της έρευνα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να ε, μπορέσει να βάλει στο περιθώριο την χρηματοδότηση της οικονομίας και να προωθήσει την χρηματοδότηση της ε, οικονομίας. Κερδίζει προσπάθειες των χωρών μελών να για την ολοκλήρωση του ενοποίηση του προπολογισμού. Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στο διοικητικό έλεγχο Σύμφωνα με την χώρα πολιτική των χρωρών μελών, με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να υπάρξει μια υγιής διαχείριση. Τρίτον, το Συμβούλιο πρότεινε να αφήσει απρεκή περιθώρια κάτω από τα νότατα όρια του, του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου για να μπορέσει να αντιμετωπίσει απρόβλεπτες καταστάσεις. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, θα επιθυμούσα τώρα να αναφερθώ στα βασικά στοιχεία της άποψης του Συμφουλίου όσον αφορά τα διάφορα κονδύλια και υποκονδύλια του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου. Ξεκινώντας από την ευφυή ε, και ολοκληρωμένη ανάπτυξη, το Συμβούλιο αποδίδει μεγάλη σημασία στο κεφάλαιο αυτό γιατί αντιστοιχεί σε ένα τομέα που δράσει τη Ευρωπαϊκής Ένωση ιδιαίτερη προστιθέμενης αξίας διαταματίζοντα ένα κομβικό ρόλο στα πλαίσια τη στρατηγικής Ευρώπης 2020 ιδιαίτερα στον τομέα της έρευνας, της ανταγωνιστικότητας, της επιχειρηματικότητα και τη καινοτομία υπό το κεφάλαιο ε, έννοια η ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη και εργασία στο Συμβούλιο υποστηρίζει τις δράσεις που είναι υπέρ της ανταγωνιστικότητας και ιδιαίτερα αυτής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και για επενδύσεις στον τομέα της παιδείας, των ανθρωπίνων δεξιοτήτων και στο Εράσμους για όλα τα προγράμματα. Οι μειώσεις που, οι μειώσεις που αφορούν αυτό το κεφάλαιο αφορούν μεγάλα προγράμματα υποδομών και αυτό βασίζεται σε, στις αναμενόμενες δυνατότητες απορρόφησης. Αλλά υπάρχει το θέμα της συμπλήρωσης των προηγούμενων προγραμμάτων. Η μείωση που εφαρμόζεται από το Συμβούλιο σε μεγάλα προγράμματα όπως για παράδειγμα το ΙΤΕΡ e e και το Trans, τα ευρωπαϊκά δίκτυα είναι ευθυγραμμισμένο με την προσέγγιση που πρόσφατα πρότεινε η Επιτροπή για να μπορέσουν να αυξηθούν τα κονδύλια για το Horizon 2020, Εράζους και ε, Κόσμες για τα πρώτα χρόνια του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου και για να μπορέσει να αντισταθμιστεί αυτό αναβάλλοντας ορισμένες δαπάνες για τα επόμενα χρόνια. Το Συμβούλιο κατέβαλε μια προσπάθεια να διασφαλίσει ένα παρκέ επίπεδο πληρωμών για διαθροτικές δράσεις. Συνεπώ αποφάσισε ότι υπό το 1 δι αυτά, δηλαδή οικονομική, κοινωνική και δαφική συνοχή, θα πρέπει να υπάρξει μια αύξηση των πληρωμών κατά 7,5% ε, σε σύγκριση με το 2013. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τη 27ης και 28ης Ιουνίου, η πληρωμή 6 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ε, πρωτοβουλία που αφορά την νεολαία ε, αφορά ε, δικαιούχου σε περιοχέ που πλήττονται από υψηλά επίπεδα ανεργία των νέων και αυτό θα ξεκινήσει από τον Ιανουάριο του 2014. Σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο 2, βιώσιμη ανάπτυξη και φυσική πόρη, το Συμβούλιο προτείνει να σταθεροποιήσει το επίπεδο των πληρωμών σε σχέση με το 2013. Παρόλα ε, ή των δεσμεύσεων ε, ε, συμφωνεί να αυξήσει τις δεσμεύσεις για δαπάνες που έχουν σχέση με την αγορά και άμεσες πληρωμές στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εγγύσεων κατά 0,28%. Η μείωση σε αυτό το κεφάλαιο κατανέμεται μεταξύ του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου για Γεωργική Ανάπτυξη και τα, το, το, τα, Ταμείο Πόρων. Με βάση τις ε, τελευταίες πληροφορίες που έχουμε ε, στη διάθεσή μας και που μπορούν να θεωρηθούν μετά από την παρουσίαση από την Επιτροπή. Σε ό,τι αφορά το σημείο 3, ασφάλεια και υπηκότητα, ε, εκεί ε, το Συμβούλιο θεωρεί ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ρεαλιστικές δυνατότητες απορρόφησης. Σε ε, ε, ό,τι αφορά τις δαπάνε, το Συμβούλιο συμφωνεί με την Επιτροπή σε ό,τι αφορά το θέμα του ασύλου και της μετανάστευση και τι συναφείς πρωτοβουλίε που αφορούν τα εξωτερικά σύνορα, τη δικαιοσύνη, εσωτερική ασφάλεια, προστασία του καταναλωτή και δημόσια υγεία. Σε ό,τι αφορά το 4, Global Europe, το Συμβούλιο θέτει ε, τις ε, δεσμεύσεις και τις πληρωμές σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό που προτείνεται από την Επιτροπή για να μπορέσει να αντικατοπτρίζει καλύτερα τις εφαρμογές του προπολογισμού και για να ληφθούν υπόψη δυνατότητες απορρόφησης. Αυτό το σημείο μαζί με τα σημεία 1α και 1β και καθώς και το 2 υπόκεινται σε μία δήλωση που αφορά τις δεσμεύσεις πληρωμών, οι οποίες το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ένα σχέδιο προϋπολογισμού με δεσμεύσεις πληρωμών για το 2, αν οι δεσμεύσεις πληρωμών είναι ανεπαρκείς για να καλύψουν τις δαπάνες υπό αυτά τα προβλέπονται σε αυτά τα κεφάλαια. Σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο 5, διοίκηση, το Συμβούλιο αναγνωρίζει τι προσπάθειε που κατεβλήθησαν από τα θεσμικά όργανα για να περιοριστεί η αύξηση στι ε, υπολογισμού του προπολογισμού συμπεριλαμβανομένη και τη μείωση του αριθμού του προσωπικού, σύμφωνα με το στόχο του 5% το χρονικό διάστημα 2015 4-17. Παρό, ε, ε, ε, πέραν αυτού εντοπίστηκαν και άλλες δυνατότητες να γίνουν οικονομίες. Το Συμβούλιο προτείνει να εξαλειφθούν οι δεσμεύσεις που συμπεριλαμβάνουν προσαρμογές μισθών το 2011 και το 2012. Το Συμβούλιο θεωρεί ότι αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να προδικάζεται η απόφαση του, ε, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Το Συμβούλιο υποστηρίζει συγκρίσιμε μειώσεις και, στον τομέα, και στις δεμεύσεις και στις πληρωμές ανάλογα με τον αριθμό του προσωπικού και η αυτοχρηματοδότηση γίνεται αποδεκτή. Το Συμβούλιο συνήθως δεν τροποποίησε το τμήμα του προπολογισμού που αφορά το Κοινοβούλιο. Τέλο, σε ό,τι αφορά το σημείο 6, το Συμβούλιο συμφωνεί με το επίπεδο των δεσμεύσεων που προτείνονται από την Επιτροπή. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, Είμαι όσο ότι η θέση του Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο προπολογισμού 2014 αντιπροσωπεύει, αποτελεί μια εξισορρόπηση μεταξύ της ανάγκης του να συνυπολογίσουμε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση στις χώρες μέλη και της ανάγκης να διασφαλίσουμε επαρκείς δεσμεύσεις στο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουμε να στηρίξουμε νέα προγράμματα και δράσεις προωθώντα την ανάπτυξη και ε, την ε, εξέλιξη. Όλοι μας ε, συμφωνούμε για την σημασία και προστιθέμενη αξία προγραμμάτων και δράσεων ε, που αναπτύσσονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όλοι υποστηρίζουμε ότι θα πρέπει να χρηματοδοτούνται ανάλογα, όπως το κάνουν και οι Υπουργοί Οικονομικών. Όλοι μας όμως δεσμευόμαστε από τους στόχους ε, της δημοσιονομικής επιθαρχίας και τις προσπάθειες που κάνουμε να μειώσουμε τα ελλείμματα. Κάθε επιπλέον ευρώ στην προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάζει τους εθνικούς προπολογισμούς. Αυτό είναι μια δέσμευση που μας αφορά όλους. Κατά συνέπεια, όλοι μας θα πρέπει να θέσουμε προτεραιότητες και να βρούμε τις σωστές ισορροπίες, διασφαλίζοντας από τη μία φορά την έγκαιρη εφαρμογή των προγραμμάτων και δράσεων και από την άλλη πλευρά περιορίζοντας τα ελλείμματα στους εθνικούς προπολογισμούς στα πετούμενα επίπεδα. Βασίζομαι στη δική σας κατανόηση και στη δική σας στήριξη σε ό,τι αφορά τα παραπάνω θέματα. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το δημοσιονομικό έτο 2014 θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη τη οικονομία επενεργώντα ως καταλήτη για ανάπτυξη και ε, εργασίες ε, αλλά και στο επίπεδο μόχλευσης. Ελπίζω ότι ο κοινό αυτός στόχος θα, οδηγήσει, θα καθοδηγήσει όλους μας κατά τη διάρκεια των συζητήσεων τους επόμενους μήνες από τη στιγμή που είναι στόχος όλων μας η επίτευξη συμφωνίας για τον προπολογισμό του 2014. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Mr. Ε, Rimkusas, I give the floor to Mr. Lewandowski. President, Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ, ε, Σήμερα η σημερινή συνεδρίαση είναι η δεύτερη ευκαιρία που έχω μετά τον τριμερή διάλογο να εκφράσω τη βαθύτατη ανησυχία μου με την ανάγνωση του προπολογισμού του 2014 από το Συμβούλιο. Παρουσιάζοντα το σχέδιο για το 2014 η Επιτροπή είχε ένα ξεκάθαρο μήνυμα δεν μπορούμε να προσποιηθούμε ότι τα πράγματα παραμένουν ως είχαν για πολλούς λόγους αυτό το οποίο γίνεται, γίνεται μέσα σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο, πιο αργά από τη συνήθως, από τον Ιούνιο, για να έχουμε ένα σταθερό πλαίσιο για το σχέδιο προϋπολογισμού. Στην πρότασή μας, λόγω των χαμηλών ορίων για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές, ε, η πρότασή μας ε, ήταν μείωση των δεσμεύσεων κατά 6%, 9,1 δις λιγότερα δηλαδή από αυτά τα οποία χρειαζόμαστε για φέτος και για τις πληρωμές 8,4 δις λιγότερα από αυτά που χρειαστήκαμε το 2013. Επομένως δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι κάνουμε περικοπές ως συνήθως και γι' αυτό ακριβώς ανησυχούμε με την ανάγνωση του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο ακολουθεί τον παραδοσιακό τρόπο περικοπών στην αναγνωσή του, αλλά εδώ είμαστε ήδη σε πολύ χαμηλό επίπεδο για το 2013. Περικόπτουν οι δαπάνε κατά 240 ε, ε, ε, εκατομμύρια πράγμα το οποίο είναι ε, υπερβολικό. Ε, δεν μπορώ να παρακολουθήσω το σκεπτικό του Συμβουλίου, γιατί γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να ενισχύσουμε την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη, που έχουμε μια μικρή ανάκαμψη φέτος και ελπίζουμε να τονωθεί του χρόνου. Ξέρουμε ότι η χρηματοδότηση των διαθωτικών των διαθρώσεων είναι ένας τρόπος πρόθεσης της ανάπτυξης και τις κύριες περικοπές της χρηματοδότησης το Συμβούλιο της κάνει στον τίτλο που προτείνει ε, το κόσμο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το πρόγραμμα Horizon 2020 ε, για τόνωση των, της πρωτοβουλίας. Ε, αυτές, αυτές λοιπόν οι περικοπές του Συμβουλίου θα προβούν εις βάρος ε, της ανάπτυξης. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας αυτά τα οποία συμβαίνουν και γύρω από την Ευρώπη. Στη Συρία παραδείγματος χάρη, για να λάβουμε υπόψη μας ε, όλα αυτά τα οποία σημαίνουν υποχρεώσεις μας και προς τον εξωτερικό κόσμο. Δεν μπορώ να δεχθώ τις δικαιολογίες του Συμβουλίου ότι αυτό γίνεται γιατί χρειαζόμαστε ένα περιθώριο ευελιξίας για κάποιες απρόσμενες εξελίξεις το 2014 διότι ε, μέσα στο, στα όργανα τα οποία έχουμε υπάρχει δυνατότητα κινητοποίησης μέσων ευελιξίας μέσα στα περιθώρια τα οποία δίνονται. Δεν μπορούμε να κάνουμε παραπάνω περικοπές για να έχουμε περιθώριο. Αυτό συμπεριλαμβάνεται το να συνεχίσουν να μειώνουν κάτι το οποίο έχει ήδη μειωθεί θα καταλήξει στο να μην ανταποκρίνεται στις ανάγκες του 2014 και αυτό είναι ανησυχητικό. Ξέρουμε ότι υπάρχει ε, ο κύκλος ζωής των προγραμμάτων ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν τελειώνει το 2013. Υπάρχει το νησιν και έχουμε ε, τη συνέχιση των προγραμμάτων το 2014. Ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση στην αγορά εργασίας στην Ευρώπη. Και επομένως πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε αυτή τη φορά μια προσπάθεια και ίσως η κνήμα συνάντηση σχετικά με τις πληρωμές μπορεί να αποτελέσει μια ευκαιρία για να συζητήσουμε τις εξελίξεις στις πληρωμές και να δούμε ε, κατά πόσο έχουν οριμάσει τα μεγάλα προγράμματα στην Ευρώπη και πώς εξελίσσεται η ορίμανση των προγραμμάτων και ελπίζω ότι αυτή θα είναι μια ευκαιρία να συζητήσουμε μια λογική προσέγγιση στον προϋπολογισμό σε αυτή την κρίσιμη στιγμή της ευάλωτης ανάκαμψης στην Ευρώπη. Ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός είναι πολύ ε, ειδικό γιατί το 90% των πιστώσεων ε, είναι είτε μη διαφοροποιημένες ε, δαπάνες και μόνο το 10% αφορά νέα προγράμματα για την ε, νέα περίοδο 2014-2020. Αν το δικαστήριο ε, καταλήξει μια διαφορετική απόφαση θα μπορούσαμε να προσαρμοστούμε αντιστοίχως και όχι εκ των προτέρων. Και η Διοργανική Συμφωνία λέει ότι όλα τα θεσμικά όργανα είναι υποχρεωμένα να επιδιώξουν μείωση κατά 1% και κανένα θεσμικό όργανο δεν απαλλάσσεται από αυτή την υποχρέωση. Ζητώ λοιπόν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αξιότιμοι κυρίε και κύριοι βουλευτέ, να λάβει υπόψη αυτά τα επιχειρήματα όταν προετοιμάζετε την ανάγνωσή σα για τον προπολογισμό του 2014. Σας ευχαριστώ για τις προσπάθειές σας να προετοιμάσετε εγκαίρως ε, τις προπαρασκευαστικές δράσεις, τον κατάλογο με τις προπαρασκευαστικές δράσεις και ελπίζω ότι θα έχουμε πολύ καλή συνεργασία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του προϋπολογισμού. Τώρα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτά τα οποία ε, τώρα είναι η γνώση μας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ε, και η συμφωνία τελευταία στιγμή για το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο σχετικά με το front loading ή το back loading, αλλά κυρίω το front loading για το κόσμο και το Εράσμους. Θα πρέπει η δεύτερη ε, τροποποιητική επιστολή να είναι πολύ συγκεκριμένη για τη Γεωργία και την Αλία. Ας είμαστε αισιόδοξοι ότι θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε μέσα σε 21 μέρες ε, το έργο μας κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης και ελπίζω να είναι καλό το αποτέλεσμα των ε, διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ. ευχαριστούμε πολύ κύριε Βαντόφσκι. Κύριε Επίτροπε, και τώρα δώσουμε το λόγο στην κυρία Χόλμα, που είναι η εισηγήτρια. Κύριε Πρόεδρε, Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Πίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχήν για τον γενικό προϋπολογισμό, δύο-τρεις παρατηρήσεις πριν περάσω στον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου. Άκουσα και σέβομαι την άποψη του ότι αυτό που είπε η Προεδρία του Συμβουλίου ότι δεν είναι γενικές περικοπές. Έχω την εντύπωση ότι τελικά προσπαθούμε να κάνουμε περικοπές στον προϋπολογισμό για να ε, αντιμετωπίσουμε ε, τις γενικότερες ε, απαιτήσεις. Και η συνάδελφος Άννη Γένσεν φαντάζομαι θα υποστηρίξει αυτή την άποψη. Όσον αφορά τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήθελα να προσθέσω ότι καταρχήν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ε, γνωρίζει ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη κατάσταση. Αυτή η ιδιαίτερη κατάσταση ε, ε, λαμβάνει υπόψη το 2,2% ε, που είναι, ε, έχει σχέση και με την φετινή περίοδο του Κοινοβουλίου προσπαθούμε να έχουμε στενή συνεργασία με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή Περιφερειών. Μέχρι τώρα δεν έχουμε συγκεκριμένα νούμερα και υποθέτω ότι αυτά τα συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία θα τα έχουμε στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Προσπαθούμε να έχουμε ένα μείον 0,3% πέραν του κόστους της ε, νομοθετικής περίοδου και του κόστους ένταξης της ε, Κροατίας. Ε, θα ήθελα επίσης να σχολιάσω σχετικά με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Δεν είμαι σίγουρη αν το Συμβούλιο παραμένει στην απόψή του σχετικά με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. 1,7% αύξηση για ένα οργανισμό ο οποίος τώρα δημιουργείται δεν νομίζω ότι δείχνει ότι το Συμβούλιο παραμένει πιστό στη θέση του ότι θέλει να έχει αυτό τον οργανισμό. και, για, και χάρη ασφαλείας και χάρη των συζητήσεων που θα γίνουν σχετικά με τις αποκαλύψεις του Σνόντεν και την τεχνολογία, πιστεύω ότι χρειάζεται χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Παρακαλώ ε, το Συμβούλιο να λάβει υπόψη τι αναλύσει που έχουν γίνει ώστε να μπορέσει κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων να γίνει μια εμπεριστατωμένη συζήτηση. Έχω κατά κάποιο τρόπο την συζήτηση ότι ακολούθησε μια γενική πολιτική μείωση στο Συμβούλιο χωρί να λάβει υπόψη τι συγκεκριμένε περιστάσει. Θέλουμε να έχουμε ένα προπολογισμό για φέτο και προπολογισμού και για τα άλλα θεσμικά όργανα που να έχουν πραγματικό νόημα. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η άμεση αντίδραση από πλευρά Κοινοβουλίου όσον αφορά το σχέδιο του προπολογισμού είναι κάτι που χαρακτηρίζεται από απογοήτευση και ότι θα έπρεπε να υπάρξουν εγγυήσει για ανάπτυξη, για απασχόληση και αυτό θα πρέπει να εκφράζεται μέσα των πιστώσεων πληρωμών. Και ξέρουμε ότι αρχή τα όρια είναι τόσο χαμηλά που δεν μπορεί να τηρήσει τι δεσμεύσει το Κοινοβούλιο. Πρόκειται για κάτι το οποίο είναι αφόρετο και απαράδεκτο. Και ήδη είχαμε πει ότι η Κομισιόν έχει πέσει κάτω από το 6% για φέτος. Επομένως, ε, αυτό το οποίο θέλουμε να υπάρχει κάποιος προπολογισμό βέβαια με κάποιες περικοπές, αλλά θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με καινοτομία και έρευνα το Κοινοβούλιο ε, αντίθετα με τη συμβουλία του Ιουλίου για το σε δημοσιονομικό πλαίσιο ε, κάνει περικοπές και σε αυτούς τους τομείς. Οπότε είπαμε εδώ πέρα θα πρέπει να ανέβουν το 2014 οι πιστώσεις για καινοτομία και έρευνα. Επομένως είναι ένα σκάνδαλο το ότι το Συμβούλιο πάει αντίθετα με αυτή τη συμφωνία. Θα πρέπει εμείς να κάνουμε ό,τι μπορούμε τόσο ώστε να υπάρξουν εγγυήσεις για προγράμματα, για πρωτοβουλίε, για να απασχολήσουν των νέων, για την ανάπτυξη. Γιατί σε πάρα πολλέ χώρε τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά όσον αφορά την ενεργεία των νέων. Επίση υπάρχουν κάποιε περιοχέ, κάποιοι τομεί του υπολογισμού που έχουν και άλλε περικοπέ. Ε, τώρα είπαμε ότι έχουμε ένα σωρό ε, πρόσφυγες από την ε, Συρία αλλά και εκεί θα πρέπει να υπάρχει κάποια ε, αύξηση. Έχουμε επίσης περικοπές παντού το τόσο πολύ που καθίσταται αφόρητη αυτή η πρόταση. Επίσης το ίδιο ισχύει για τις κοινωτικές περιφερειακές υπηρεσίες και κατά τη γνώμη μας οι εποπτικές αρχές όσον αφορά ε, τα χρήματα οικονομικά ε, και θα πρέπει να παρακολουθήσουν πάρα πολύ καλά την κατάσταση και να δούμε πώς οι πληρωμές θα ενταχθούν στον προπολογισμό για να μπορέσουμε να καλύψουμε τα μεγάλα προγράμματα για πολλά χρόνια. Έχουμε κάποιες περικοπές βέβαια, αλλά τα πράγματα μπαλώνονται τώρα όμως κατέβασε τόσο πολύ το τον πύχη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Δεν θα πρέπει να βρεθεί σε αυτή τη θέση το, η Επιτροπή. Επομένω, και εμείς τις επιστώσει πληρωμών, τις διαπραγματεύσει που έπονται ε, θα, τι τις προσέξουμε πάρα πολύ. είναι δύσκολε σκληρέ αυτέ οι διαπραγματεύσει και πρόκειται βέβαια να εξαρτηθούν με το τι θα γίνει με τον διορθωτικό προπολογισμό. Πάντω. από τώρα έχω να σας πω το εξή. Ευχαριστούμε τη Λιθανική Προεδρία για ε, την προπαρασκευαστική εργασία που έκανε. Ήταν καλή η συνεργασία και βέβαια όποιος ε, θέλει μπορεί. Οπότε θα πρέπει και θα προσπαθήσει να βρει λύσεις η Λιθανική Προεδρία. Αλλά ξέρω ότι είστε πολύ στριμωγμένοι γιατί πάρα πολλές χώρες ε, το μόνο το οποίο θέλουν να κάνουν είναι να κάνουν περικοπές, να κάνουν οικονομία, χωρίς να εξετάζουν τι θα γίνει στην πραγματική οικονομία. Ε, Α φροντίσει επιτέλου η Κομισιόν να τη τι δεσμεύσει τη φάσουν πάρα πολύ, κυρία Γέντσεν, λέει ο Πρόεδρο. Και τώρα. Το λόγο έχει ο κύριο Αλέλα Μασούρ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, μόνο μία φορά θέλω το λόγο όσον αφορά τον προπολογισμό του 2014 αλλά και τον ε, διορθωτικό ε, διότι και οι δύο προπολογισμοί ε, έχουν το, το, το, τον ίδιο φραγμό. Το θέμα είναι το κατά πόσον θα τηρηθεί ε, το, το, η θεσμική συμφωνία όσον αφορά το πολιτές πλαίσιο. Διότι είχαμε πει ότι θα πρέπει να υπάρχει ομοφωνία στο ανώτατο επίπεδο μεταξύ των 28. Παρ' όλα αυτά όμως ε, οι Υπουργοί των Οικονομικών αγνοούν τη συμφωνία εκείνη, την παραβιάζουν. Γιατί στις 2 ε, Σεπτεμβρίου έχουμε περικοπές ε, όσον αφορά τις προτάσεις για, τα, για τις πολιτικές προτεραιότητες, τις προτάσεις της Τα είπε η Επιτροπή μας, τα είπε ο εισηγητής όσον αφορά τις ΜΜΕ, το έρασμος για όλους, όσον αφορά τα ιδιωτικά ταμεία, όλα όσα οθούν στην ανάπτυξη. Επομένως, τι ωφελεί, τι εξυπηρετεί η Κορεπέρα, εάν δεν είναι δυνατόν δεν μπορεί να ενημερώσει τους υπουργούς οικονομικών σε σχέση με τις αποφάσεις που έχει βουλευτεί από το Συμβούλιο σε πολιτικό επίπεδο και που έχουν ε, επίσης ε, επικυρωθεί σαν αποφάσεις από το, από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Επομένως θα πρέπει να, να υπάρχει κάποια πειθαρχία σε αυτό που αποφασίζονται από του υπουργού. Ε, εδώ, Πολλού μήνες συζητήσαμε για το πολιτές πλαίσιο και τον ε, Ιούλιο με ευρία πλειοψηφία εγκρίθηκε η συμφωνία από το Κοινοβούλιο. Επομένω ήρθε η ώρα όλοι να επιδείξουν καλή πίστη, να ε, τιμήσουν αυτές τους τις δεσμεύσεις που ήταν επισήμως ε, αν είχαμε πει ότι αν δεν συμφωνούμε σε όλα δεν υπάρχει συμφωνία σε τίποτα. Εξευρέθηκε όμως σημείο συμφωνία ε, για όλα. Επομένως τώρα θα πρέπει να, να ανατηρηθεί η συμφωνία. Πάκτα σουν σερβάντα. Θα πρέπει τα, τα συμπεφωνημένα να, να, να, Και για, το, ε, και για το και για το 2014. τώρα έχουμε βρεθεί τώρα να υπάρχει έλλειμμα όσον αφορά την πρώτη δόση και είπαμε να πάμε στο, στα, στα 3 της 900 αλλά όσο δεν υπάρχει επίσης συμφωνία για αυτή την ε, δόση ε, όσο κάποια αρμόδια και το ε, υπηρεσία Συμβουλίου δεν έχει δώσει το πράσινο φως τότε η κύρωση του πλαισίου 2014-2020 δεν πρόκειται να κατέβει σε ψήφιση για την όλη του Κοινοβουλίου. Είχε προβλεφθεί για το πολιτέ πλαίσιο να γίνει σε αυτή την ε, σύνοδο η ψήφιση. Αυτό πρόκειται να γίνει αύριο. Τώρα όμως αυτό αναβλήθηκε για την ε, δύο μήνες πιο μετά για τη δεύτερη ολομέλεια του, του Οκτωβρίου. Όμως, ε, και θα και το αεροκόρμη και άλλο να χρειαστεί. Ε, έχουμε ε, κάνει, είπαμε, μια, έναν τριμερή διάλογο, ευχαριστώ την Προεδρία, συνέχιση το ρεκόρμη της Προεδρίας και μόνος έτσι μας σε αυτή την βάση θέλουμε να ρυθμίσουμε τα θέματα του τρέχουσας κρίσης του 2014 γιατί γίνανε όλες οι πολιτικές κινήσεις, όμως τώρα θα πρέπει όλα αυτά να υλοποιηθούν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λαμασούλη, ο Πρόεδρος. Και τώρα θα δώσω τον λόγο και πάλι στον κύριο Ριμκούνας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο κύριο Λεβαντόφσκι, την συγγήτρια Χολμάιερ και Γιάννησεν και τον πρόεδρο τη Επιτροπή Προπολογισμών, κύριο Λαμασούρ, για τι ε, πολύ χρήσιμε παρατηρήσει του. Αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι η καλύτερη κατανόηση των θέσεών μας και των θέσεων της Επιτροπής σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου είναι ο βασικός μας στόχος και νομίζω ότι προχωρούμε και ανοίγει για μας η πόρτα για να ξεκινήσουμε τις πραγματικές διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό του 2014 κατά τους επόμενους μήνες. Θεωρώ ότι η σημερινή συζήτηση ήταν μια πολύ καλή αφετηρία και θα προχωρήσουμε. Εμείς βασιζόμαστε στην υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πάντοτε η Επιτροπή παίζει το ρόλο του έντιμου και ικανού μεσάζοντα και ευχαριστούμε τον Γιάννου Λεβαντόφσκι για την καλή του συνεργασία. Σας διαβεβαιώνω ότι η Λιθουανική Προεδρία του Συμβουλίου και εγώ ίδιος θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να επιτύχουμε θετικά αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Και εύχομαι κάθε επιτυχία στο Κοινοβούλιο όταν θα εξετάζετε τη θέση του Συμβουλίου τις επόμενες εβδομάδες και περιμένουμε τη συνεργασία μας κατά τον Οκτώβριο και Νοέμβριο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πέρα τη συζήτηση. Περνάμε τώρα στην έκθεση Λαβία. Σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού